Άρχεται λοιπόν η συνεδρίαση και θα ξεκινήσουμε με τα κείμενα τα οποία εγκρίθηκαν χθε και τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης. Εάν δεν υπάρχουν ε, παρατηρήσεις, θεωρούνται εγκεκριμένα.